πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τους ιδίους πόρους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Υπάρχει κατάλογος ομιλητών. Πρώτος θα είναι ο κύριος Αρτουή, Πρόεδρος Επιτροπής Προπολογισμών για τρία λεπτά παρακαλώ. Διαδικαστικό. Sorry, Αυτό το αίτημα κατεπήγοντος μου δημιουργεί τρεις απορίες. Πρώτον, για τρεις εβδομάδες, οπότε και είχαμε τη διαδικασία συνδιαλλαγής για το σχέδιο του προϋπολογισμού 2015 και για τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς ε, του 2014, το Συμβούλιο κινητοποιήθηκε, έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον τόσο πολύ που τοποθετήθηκε για τη συνδιαλλαγή λίγες ωρίτσες πριν λήξει όλη αυτή η προθεσμία. Και έτσι βέβαια απέτυχε η συνδιαλλαγή. Και πραγματικά ε, φαίνεται ότι τους άφησε εξαντλημένους στο Συμβούλιο η ανασχόλησή τους με αυτό το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, λόγω ακριβώς της αποτυχίας, προτείνει 420 εκατομμύρια επιπλέον πόρους σε σχέση με τα στελωνιακούς δασμούς και κάποια άλλους φόρους και τέλη, όχι για να ε, συμβάλλει στην τακτοποίηση των ανεξόφυτων λογαριασμών και ποσών, αλλά για επιστροφή αυτών των χρημάτων στα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να πω ότι με τον τρόπο αυτό και σε αυτό το θέμα από τη μία έχουμε την αναδρομική ισχύ και από την άλλη έχουμε το κατεπήγον. Πρέπει να κάνουμε μια επιλογή. Εμείς αποφασίσαμε αναδρομική ισχύει αναδρομικότητα, άρα δεν υπάρχει λόγος να βιαζόμαστε αποφασισαμε αναδρομικη ισχυ αναδρομικοτητα πολύ. Αυτές είναι οι απορίες μου και ήθελα να τις ε, μεταφέρω και στους αξιότιμους βουλευτές. Thank you. ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τώρα δύο συνεισηγητές, οι οποίοι θέλουν το λόγο. Συνάδελφοι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Με συγχωρείτε, δεν σας είδα, δεν σας άκουσα. Έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν μπορεί οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να φτάσουν εδώ. Υπάρχει μποτιλιάρισμα τρομερό. Υπάρχουν κάποιοι που λείπουν, ε, όμως χωρίς να το θέλουν διότι λόγω της επίσκεψης του Πάπα δεν, κινείται, δεν κινούνται τα αυτοκίνητα. Αυτό είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Παρακαλώ να το λάβετε υπόψη ως διαδικαστικό. Δεν μπορούμε να φτάσουμε εδώ παρότι θέλουμε να είμαστε εδώ εγκαίρως. Σας ευχαριστώ πολύ για την επισήμανση. Είναι αρκετοί συνάδελφοι όμως μέσα στην Όλο μέλη αυτή τη στιγμή. Πάντως σημειώνω την παρατήρησή σας. Κύριε Τεραμπερά, διαδικαστικό. Ναι, Πρόεδρε, θέλω απλώ να σα καθησυχάσω και να διαβεβαιώσω ότι οι σοσιαλιστέ και οι δημοκράτε δεν ε, κοιμούνται περισσότερο από του άλλου, δεν είναι υπναράδε. Ο Ματέο Ρέτσι είναι σε συνεδρίαση μαζί του. Θα έρθουν όλοι μαζί. Είναι τώρα όλοι μαζί σε μια συνεδρίαση και θα καταφτάσουν. Σα ευχαριστώ για του για, για τους λέει η πρόεδρο. Θα συνεχίσουμε. Έχουμε δύο συνεισηγητέ. Δίνω το λόγο για 1,5 λεπτό πρώτα στον κύριο Ντεπρέ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το Συμβούλιο στα κατεπίγοντα χαρακτήρα για να επιτρέψει ορισμένα κράτη-μέλη να πραγματοποιήσουν πληρωμέ που έπρεπε να έχουν από την 1η Δεκεμβρίου αναπτύξει στον προπολογισμό τη Ένωση, που ήδη είχαν ορίσει. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν υπάρχει κατεπίγουσα ανάγκη αυτή τη στιγμή να χορηγηθούν μεγάλα ποσά σε ορισμένα κράτη-μέλη ακόμη και αν για, αυτά, για ορισμένα από αυτά φανεί πικρό το χάπι. Εδώ έχουμε να κάνουμε έναν διορθωτικό προπολογισμό, ένα προπολογισμό για το 2015 που θα επιτρέψει να τιμηθούν οι δεσμεύσει και οι υποχρεώσει που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ίδια. Το κατεπίγον σήμερα είναι να εγκριθούν οι διορθωτικοί προπολογισμοί του 2014. Αυτό είναι απαραίτητο για να σταθεροποιηθεί. Σημειώνω σταθεροποιηθεί και όχι να περιοριστεί το ποσό ποσό των ανεξόφλητων λογαριασμών που θα φτάσει έτσι στα 30 δις ευρώ στο τέλος του έτους. Κατεπήγον είναι σήμερα να συμφωνήσουμε σε ένα πολιετές οικονομικό σε ένα πολιετέ πλαίσιο για σταδιακή εξόφληση των ανεξόφλητων, ώστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα τη αφαιρεγκαιότητα τη Ένωση, είτε λοιπόν με ε, την ε, ορθή εξόφληση είτε με απαράδεκτες και αφόρητες καθυστερήσεις εξοφλήσεων των λογαριασμών. Το αίτημα του Συμβουλίου δεν έχει καμία βάση ή αιτιολογία. Το να αποδώσουμε αυτή, να αναγνωρίσουμε αυτό το κατεπήγοντα χαρακτήρα θα σήμαινε ότι δίνουμε δίκιο στο Συμβούλιο το οποίο ομφαλοσκοπία ασχολείται με τα εσωτερικά του προβλήματα και δεν τιμά τις δεσμεύσεις του. Ευχαριστώ. Κύριε Λεβαντόφσκι, εσείς ως συνεισηγητής μισή λεπτό. Θέλω να συμπληρώσω ορισμένα πράγματα στα όσα είπε ο συνάδελφος και να δώσω λίγο το πλαίσιο και το υπόβαθρο του αιτήματο αυτού για τον κανονισμό των ιδιών πόρων στο τέταρτο, τέταρτη τροπολογία. Το Κοινοβούλιο σημειώνει ότι κατεπίγουσα ανάγκη είναι να ε, καλυφθούν οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί και ω εκ τούτου να τιμηθούν οι υποχρεώσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά την απόφαση για του ιδίου πόρου, επρόκειτο για μια απόφαση ομόφωνη των κρατών μελών, αποφασίστηκε από τα κράτη-μέλη. Έχουν ε, ε, γίνει αναθεωρήσει οι οποίες συνεπάγονται τώρα την επιστροφή σε ορισμένα κράτη ποσών και την επιπλέον καταβολή από ορισμένα κράτη ποσών, αλλά αυτό σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το παράδοξο λοιπόν είναι ότι εμεί ζητούμε κατεπίγουσα ανάγκη για ορισμένε χώρε, μία-δύο χρόνια και ευελιξία, χώρε όμω οι οποίε δεν ήταν ποτέ ευέλικτε και του αντίον βραδιμπορούσαν και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να καθυστερήσουν την επίλυση των προβλημάτων στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Είμαστε διατεθειμένοι με να το κάνουμε αυτό, αλλά όχι με διαδικασίε κατεπίγουσε. Μέσα σε ένα χρονικό σε ένα λογικό χρονικό πλαίσιο και με ε, ταυτόχρονη εξόφληση των υποχρεώσεών μας, το να τιμούμε ως Ένωση, ως Κοινοβούλιο, ε, τους λογαριασμούς μας προς επιχειρήσεις, προς ιδιώτες και φορείς, είναι ζήτημα αξιοπρέπειας και αξιοπιστίας ημών, αλλά και της Ένωσης γενικότερα. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ακούσατε τους δύο συνεισηγητές. Υπάρχει κανείς που θέλει να υποστηρίξει το αίτημα του Συμβουλίου, παρακαλώ. Δεν βλέπω να ζητεί κανείς το λόγο. Και έτσι... Το αίτημα για κατεπίγουσα διαδικασία ψηφίζεται. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. The Επόμενο θέμα στην Θα σας παρακαλέσω. Θα σας παρακαλέσω γιατί εδώ γίνεται συνεχίστη συζήτηση. Όποιος θέλει να αποχωρήσει, να αποχωρήσει ησυχώς και με σεβασμό στη διαδικασία της συζήτησης που συνεχίζεται. Έχουμε λοιπόν προφορική ερώτηση προς το ε, Συμβούλιο και την Επιτροπή για την Απασχόληση και τις Κοινωνικές Στρατηγικέ Στρατηγικές ε, Ευρωπαϊκή Ένωση 2020. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινώ τη συζήτηση δίνοντας το λόγο στην κυρία Σόγκο. Για πέντε λεπτά έχετε το λόγο παρακαλώ. Yes, you have the floor. I...